παρακαλώ να καθίσετε. Επαναρχίζει η συνεδρίαση της Ολομέλειας. Αποτελέσματα της ε, ψηφοφορίας για τους κοσμήτωρες. Παρακαλώ καθίστε και ακούστε. 684 ψήφοι. 15 άκυρα ψηφοδέλτια. Έγκυρα. 669 ψηφοδέλτια. Η απόλυτη πλειοψηφία κατά συνέπεια, η οποία είναι απαραίτητη στον πρώτο γύρο, 335 ψήφοι. Αποτελέσματα. Κυρία Γκέργερ Ντέτεμπεργκ, 237 ψήφοι. Higgins, 284. Λιμπεράσκι, Λιμπεράτσκι 222. Λούλινγκ 297. Μαστάλκα 232. Νιούτον Ντάν 177. Σπερόνι, 106. Κανένας επομένως υποψήφιος δεν συνέλεξε την απόλυτη πλειοψηφία των, ε, ψήφων, των εγκύρων ψήφων. Επομένως, δεν έχει καταληφθεί καμία θέση κοσμήτωρος και είναι απαραίτητο και ένας δεύτερος γύρος ψηφοφορίες για τους κοσμήτωρες. Θεωρώ ότι θέλουν να συνεχίσουν ως υποψήφοι όλοι αυτοί οι οποίοι είναι υποψήφοι για το αξίωμα των κοσμητών. Θέλει κάποιος να αποσυρθεί. Ως υποψήφιος, όχι. Επομένως, συνεχίζουμε στον δεύτερο γύρο με τους 7 αυτούς υποψηφίους. Σας προτείνω και αυτός ο δεύτερος γύρος να γίνει με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Machen wir das jetzt oder um 5 Uhr? Now? Now. Now. Σας παρακαλώ να καθίσετε λοιπόν και ζητώ και πάλι την προσοχή σας γιατί είναι λίγο μπερδεμένο το θέμα. Θα κάνουμε μια δοκιμαστική ψηφοφορία πρώτα. Παρακαλώ. Ε, κάνουμε μια δοκιμαστική ηλεκτρονική ψηφοφορία. και θα ήθελα να ευχαριστεί και... λοιπόν, μπορείτε να ψηφίσετε για τον Πλάσιο Ντομίνγκο, τη Χούλια Μιγένε, το... τη Μοντσεράτ Καμπαγέρ, ακόμα και τον Παβαρότη, αν και έχει αποσυρθεί μάλλον από το αξίωμα αυτό εδώ και πολύ καιρό. Λοιπόν, παρακαλώ ξεκινήστε τις μηχανές, τα τα συστήματα ψηφοφορίας. Πατάτε το κάτω ε, δεξί κουμπί. Το κάτω κουμπί λοιπόν. Και μπορείτε να βάλετε κόκκινο ή πράσινο κοντά σε κάθε όνομα υποψηφίου. Έχω γύρει κατανοητός. Μπορείτε λοιπόν να κατέβετε, να, να σαρώσετε τα, τους υποψηφίους με το κουμπί που είναι κάτω. Και μπορείτε να πείτε ναι ή όχι για κάθε υποψήφιο. Εάν δεν θέλετε να ψηφίσετε θετικά ή αρνητικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κομβίον της αποχής. Μόνο πέντε μπορούν να εκλέγουν από τους υποψηφίους. Μέχρι πέντε μπορείτε να ψηφίσετε λοιπόν. Και εάν κάνετε κάποιο λάθος μπορείτε να σβήσετε ένα υποψήφιο, να σβήσετε μάλλον τον τρόπο που ψηφίσατε για ένα υποψήφιο. Εάν λοιπόν έχετε κάνει, έχετε κάνει κάποιο λάθος, γυρίστε στον υποψήφιο και πατάτε το ακυρωτικό κομβείο και έτσι σβήνεται η ένδειξη που έχετε δώσει. Δύο φορές ναι, δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό. Λοιπόν, κάνουμε αυτή τη δοκιμασία. Καταλαβαίνετε πώς λειτουργεί το ηλεκτρονικό σύστημα ή θέλετε να θέσετε κάποιο ερώτημα. Το κάτω κουμπί είναι αυτό το οποίο σας επιτρέπει να ψηφίσετε για κάθε υποψήφιο. Συν είναι υπέρ, πλην κατά και υπάρχει και η αποχή. Μοντσεράτ Καμπαγέ, άρχεται η ψηφοφορία. ich habe gesagt, ich erkläre das für eröffnet. Άρχισε η ψηφοφορία, σας το υπενθυμίζω. Έχει αρχίσει. muss ich die Technik fragen. Εάν υπάρχει πρόβλημα και δεν έχει αρχίσει η ψηφοφορία, πρέπει να ζητήσω από τους τεχνικούς την αρρωγή τους. Yeah, bitte, Herr Κύριε Γκέμπελς, άρχεται η ψηφοφορία. Μπορείτε τώρα να ψηφίσετε. Funktionieren alle Abstimmmaschinen. Λειτουργούν όλα τα μηχανήματα. Ναι, Ihre Abstimmmaschine funktionieren nicht. Ποιανού το μηχάνημα δεν λειτουργεί. Παρακαλώ. Κύριε Μαρινέσκου. Πείτε, Μαρινέσκου. I can vote only two persons. Εγώ μπορώ να ψηφίσω μόνο δύο. This is, this is valid for the... Είναι για το τεστ μόνο. Ωραία. Yeah, das ist nur ein test. Μα μόνο μια δοκιμασία κάνουμε, λέει ο πρόεδρος. Δεν μπορούμε να έχουμε τόσους ε, τενόρους και σοπράνο σαν κοσμήτορες. Α, γι' αυτό κάνουμε μονάχα μια δοκιμασία. Haben Ψηφίσατε όλοι. Ακούστε με, είναι μία <laughs> δοκιμαστική ψηφοφορία. Δεν αντέχει το κοινοβούλιο τόσα αστέρια της όπερας. Το λέω για τέταρτη φορά. Λοιπόν. Κύριε Λάγκεν, είσαστε υποψήφιος. Μόνο μία Μόνο για ένα άτομο μπορώ να ψηφίσω. Αν πήγα να ψηφίσω το δεύτερο άτομο, τότε σβήνει το πρώτο. Μα είναι δοκιμασία, λέει. Είναι δοκιμαστική ψηφοφορία, λέει ο πρόεδρο. Και έχετε ψηφίσει όλοι. Εντάξει, τότε κλείνει η δοκιμαστική ψηφοφορία. Για να δούμε. So, Also ich habe die Ergebnisse. Εγώ τα έχω τα αποτέλεσμα και δεν φαίνονται στην οθόνη. Also ich kann Ihnen sagen, gewonnen hat Montserrat Caballé mit 291 Stimmen. 291 ψήφους πήρε η Montserrat Caballé. Okay. Και κέρδισε βέβαια. Γκέλ Τζόνσον δεν θα είναι μέλος της ε, ομάδας των κοσμητόρων. Και νομίζω ότι είμαστε πια έτοιμοι, κυρίες και κύριοι. Μπορούμε να περάσουμε στην ψηφοφορία. Ωραία. So, da löscht das mal, dann kommen wir jetzt zur tatsächlichen Wahl. Και τώρα ερχόμαστε στην πραγματική <clears throat> εκλογή των κοσμητόρων. Έχουμε 7 υποψήφιους και υποψήφιες, κυρία Γκέριγκερ, Δεύτερμπεργκερ, Χίκινς, Λιμπεράσκι, Λούλινγκ, Μαστάλκα, Νιούτον Ντόν και Σπερόνι. Πέντε μόνο από τους εφτά μπορείτε να εκλέξετε. Δεν είσαστε υποχρεωμένοι να ψηφίσετε και πέντε εάν δεν θέλετε. Μέχρι πέντε μπορείτε να ψηφίσετε. Λοιπόν, αν λειτουργούν όλα σωστά, θα... Όταν έχετε το κόκκινο φωτάκι κάτω από το όνομα, μπορείτε να πείτε ναι ή όχι και μπορείτε αυτό να το κάνετε μέχρι πέντε φορές. Αρχίζει λοιπόν η ψηφοφορία.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 sind So, darf ich fragen, Έχετε ψηφίσει λοιπόν τώρα όλοι. όλοι. Εφόσον έτσι φαίνεται, κλείνουμε την ψηφοφορία. Εψήφισαν 593. 297 είναι η απόλυτη πλειοψηφία και κανείς δεν πέτυχε την απόλυτη πλειοψηφία. Βλέπετε τον κατάλογο. Λούλινγκ 280, Higgins 263, ε, Γκέριγκερ 234, Μαστάλκα 226, 209, Λιμπεράσκι 200 ε, και λιγότερο οι άλλοι δύο. Επομένως χρειαζόμαστε ένα τρίτο γύρο όπου αρκεί η απλή πλειοψηφία.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 Meine Damen und Herren, da wir aber jetzt so schön gelernt haben zu wählen. Μα τώρα έχετε μάθει να ψηφίζετε τι ωραία. Οπότε η πρότασή μου είναι αντί για τις 8 να ψηφίσουμε τώρα τον τρίτο γύρο. So. So, meine Damen und Herren, ich darf dann... Λοιπόν, θέλω σας παρακαλέσω. Ξέρετε πώς γίνεται η διαδικασία, ξέρετε να περνάτε με τον κόκκινο δρομέα και να ψηφίσετε ναι, όχι ή αποχή. Εάν συνεχίζουν όλοι οι υποψήφοι και νομίζω ότι είναι όλοι παρόντες, μπορούμε να συνεχίσουμε. Υπάρχει κάποιος ο οποίος θέλει να αποσυρθεί για τον τρίτο γύρο. Εντάξει. Συνεχίζεται λοιπόν με τον τρίτο γύρο η ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Ich frage, Έχετε ψηφίσει όλοι και όλες. Υπάρχει αίθουσα κάποιος ή κάποια που δεν έχουν ψηφίσει. Όχι. Επομένως κλείνει η ψηφοφορία. Abgegebene 600 600 ψήφοι και είναι 300 η απόλυτη πλειοψηφία, δεν μας ενδιαφέρει διότι δεν χρειάζεται. Η κυρία Λούλινγκ, 273.